Ok, buongiorno a Καλή σας μέρα. Ξεκινάμε λοιπόν με τις εργασίες μας. Μεγάλη συνεδρίαση ψηφοφοριών που είχαμε. Είμαστε στο σημείο 7. Έχουμε λοιπόν το θέμα της κυρίας η εισηγήτριας, για την πρόταση κανονισμού σε σχέση με την υγεία των ζώων. 800 τροπολογίες κατατέθηκαν. Γνωμοδότηση Επιτροπής Περιβάλλοντος, Επιτροπής Αλληλείας, επίσης που κατατέθηκαν Έχουμε λοιπόν από αυτές τις δύο κοινοβουλευτικές επιτροπές 300 τροπολογίες. Προαναγγέλλεται λοιπόν μια αρκετά διεξοδική συνεδρίαση, αρκετά εκτενή συνεδρίαση. Υπάρχουν πολλές ε, ψηφοφορίες που απλουστεύονται με ομαδικές ε, ψηφοφορίες. Έτσι λοιπόν από το σύνολο αυτών των 420 τροπολογιών θα πρέπει να το ρυθμίσουμε. Θέλετε να παρέμβετε, έχετε τον... Σε ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Πρέπει να παρακαλέσω πρόεδρε, λέει η κυρία Πόλσεν, να θυμούνται όλοι πόσο πάρα πολύ περίπλοκο, απίστευτα περίπλοκο είναι αυτό το χαρτοφυλάκιο είναι ιδιαίτερα σύνθετο και περίπλοκο. Επί εβδομάδες διαπραγματευόμαστε και συζητούσαμε και συμφωνήσαμε με τις διαφορε... μεταξύ διαφορετικών κοινοβουλευτικών ομάδων όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι συμφωνούμε μέχρι τελευταίων λεπτομεριών. Όμως από την άλλη πλευρά πρέπει ο πίνακας ψηφοφορίας να χρησιμοποιηθεί όπως τον έχουμε μπροστά μας και παρακαλώ να υποστηριχθούν ε, οι ψηφοφορίες, οι συμβιβαστικές και οι ομαδικές ψηφοφορίες διότι πρόκειται για τις αρχές ε, πολιτικών αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν και ποια θέματα είναι αυτά τα οποία πρέπει να ρυθμιστούν. E Σε ευχαριστούμε λοιπόν και ξεκινάμε τώρα με την ψηφοφορία και θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν με σηκώνοντα το χέρι να ψηφίσουμε, διανατάσεως της χειρός. Αλλά όπου υπάρχει αμφιβολία θα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Όλοι οι συνάδελφοι που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν παρακαλώ να βάλουν την κάρτα τους στη μηχανή και να είναι έτοιμοι να ψηφίσουν. Στη συσκευή είσαστε έτοιμοι. Ψηφίζουμε δοκιμαστικά λοιπόν για να καταχωρηθεί ο αριθμός ψήφων. Ξεκινάμε λοιπόν τώρα. Τροπολογία 1 εισηγήτρια υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 67 Βοητσεχόφσκι υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 68 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Πάμε τώρα στην 65. Ένβη υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 149 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 150 Αγιούσο και άλλων υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 2. Επιτροπής Αλληλείας υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Υπάρχουν αμφιβολίες. 151 τώρα υπέρ. Κατά αποχές θα έλεγα απορρίφθηκε. Θα ελέγξουμε λοιπόν. Εντάξει. Έλεγχος ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 151. Άρχεται. working. Ah, it's working. Λειτουργεί η συσκευή σας. Ναι εντάξει. Κλείνει πέρας πληροφορίας. Siamo respinto. Απορρίφθηκε λοιπόν. Μάλιστα. Και πάμε τώρα στην της αλληλεία 3 υπέρ Διανατάσσεω της χειρός κατά αποχές θα έλεγα εγκρίθηκε έτσι απορρίφθηκε λέτε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά ελέγχουμε άρχεται η ψηφοφορία ψηφίζουμε την 3 άρχεται Μάλιστα, ζητώ συγγνώμη, απορρίφθηκε πράγματι. Απορρίφθηκε, ήταν σαφές. Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη. Το ίδιο τώρα, για το ίδιο, 152. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για να κερδίσουμε χρόνο. Γκίρλινγκ, ψηφίζουμε, άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας και το αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Και πάλι ηλεκτρονικά, 153, Βοητσεχόφσκι, άρχεται η ψηφοφορία, παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Και η 154 τέλος, ηλεκτρονικά πάλι, άρχεται, 154, Βοητσεχόφσκι, άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας, εγκρίθηκε. Ωραία. Και πάμε τώρα στην πρώτη ομάδα, Block A, ηλεκτρονικά, όλες αυτές τις τροπολογίες. Εντάξει, όχι, διανατάσσεως της χειρός. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκαν. Εγκρίθηκε η ομάδα Α. Ψηφίζουμε την 68, Envy, υπέρ της 68, κατά. Αποχές Να ελέγξουμε. Ωραία, ελέγχουμε. Ψηφίζουμε την 68. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε η 68. Ωραία. Μετά προχωράμε και πάμε στην 69. Ένβη πάλι. Διανατάσεως υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 157 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε μάλιστα απορρίφθηκε 70 ένβη υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε Πάμε τώρα στην 159. Σμιτ, υπέρ, Σμιτ, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε τώρα στο μπλοκ B, ομάδα Β, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε η κατηγορία αυτή. Η 71, ένβη, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 72, ένβη, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 161 τώρα, ε. Αποσύρθηκε, εντάξει, ωραία. Πάμε στο μπλοκ C. Ομάδα Γ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε το μπλοκ C. Εντάξει τώρα. Πάμε, τώρα στην 5 της αλληλείας. Διανατάσεως. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 165. Γκαρσία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Πάμε τώρα στη συνέχεια στην 171. Αγιούσο, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. Πάμε τώρα στην 75. Ένβη, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. Πάμε στην 177. Σίμψον, υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. 76 ένβη υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 70, 178 ε, μπαράτσου υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 78 ένβη υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 179 Λιούμπτσεβα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Η 181 Άλβες υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Αποχές, εντάξει, διανατάσσεως 182 Σίμψον υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Ε, να ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 182 Simpson ηλεκτρονικά για έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία. Chiusa la votazione. Respinto. Alzata di mano 180. Λοιπόν, 184. Υπερ κατά αποχές απορρίπτωται. 81 mv υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 185 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 186 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 187 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 188 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 189 <clears throat> είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 190 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 191 υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 192 υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 7 λία υπέρ. Κατά. Αποχές, δεκτή. 8 αλία υπέρ. Κατά. Αποχές, δεκτή. 6 αλία υπέρ. Κατά. Αποχές, δεκτή. Περιβάλλον 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 193, ενενήντα τρία. Γκαρσία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 195 Σίμψον υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 194 υπέρ. υπέρ επαναλαμβάνω. Κατά. Αποχές δεκτή. 197 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 196 Γκαρσία Γκουτιέρες υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε το μπλοκ δέλτα κεφαλαίο υπέρ κατά αποχές δεκτό. Τώρα περνάμε στην ένα ενοποιημένη υπέρ κατά αποχές δεκτή. Περνάμε τώρα στο άρθρο 6 και ψηφίζουμε την ενοποιημένη 2. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Περνάμε στο άρθρο 7 και στην ενοποιημένη 3. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συνεχίζουμε με την ενοποιημένη 4. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Ψηφίζουμε τώρα την ενοποιημένη 5. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Περνάμε τώρα την ομάδα τροπολογιών αγγλικό G ηλεκτρονική ψηφοφορία J μάλλον, J στο κείμενο για την πυκνότητα της παραγωγής. Υπάρχει σύγχυση στα αγγλικά για κάποιους βουλευτές ανάμεσα στο J και στο G. Λοιπόν. Το J λοιπόν ψηφίζουμε, το J. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Κυρία Πάουλσον, την ομάδα J ψηφίζεται. Ψηφίσατε όλοι. Απορρίπτεται. Allora, dobbiamo ripetere, scusate un attimo colleghi. Ζητώ συγγνώμη συνάδελφοι, λέει ο Πρόεδρος, ζητώ συγγνώμη. Πρέπει να επαναληφθεί η ψηφοφορία για την ομάδα αγγλικά J γιατί δημιουργήθηκαν κάποιες, ε, κάποιοι προβληματισμοί. Μετά από την ενωμένη 5, ενωποιημένη 5, μιλάμε για την ε, J συμβιβαστική. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, τέλος της ψηφοφορίας. Απερίφθη ακόμα πιο ξεκάθαρα, είχε απορριφθεί και πριν, απερίφθη για μια ακόμη φορά. Περνάμε λοιπόν τώρα στην ενοποιημένη υπαριθμών 6 επί του άρθρου 10 Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Αμέσως μετά περνάμε στην ενοποιημένη 7. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Περνάμε στην 8, στο άρθρο 12, ποιοι είναι υπέρ της ενοποιημένης 8, υπέρ κατά δεκτή. Ψηφίζουμε τώρα τη συμβιβαστική 1 του εισηγητή. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές δεκτή. Τώρα θα ψηφίσουμε την 326 του εισηγητή. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Αμέσως μετά περνάμε στην ενοποιημένη 9. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Αμέσως μετά περνάμε στην τροπολογία 352 γέγγελ του άρθρου 14. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τώρα 353 μπαράτσου ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Ψηφίζουμε την 136 Επιτροπή Περιβάλλοντος υπέρ. Κατά Θα γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος για την 136 περιβάλλον. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απερίφθη. Τώρα 3.55. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 3.56 τώρα Νταντέν ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 357 γκίρλινγκ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 358 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 33 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. 34. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 35. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συγγνώμη, ξεχάσαμε μία τροπολογία, πρόκειται για την 363. Ποιοι είναι υπέρ της 363, κατά, αποχές δεκτή. 365 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 366 γκίρλινγκ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 369 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεκτή, λάθος λέει ο πρόεδρος. Γίνεται δεκτή. Περνάμε τώρα στην 370 υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, Αποχές απορρίπτεται. 371. Συγγνώμη, 372 διορθώνει ο πρόεδρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 373. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 139. Υπέρ. κατά απορρίπτεται 39 ποιοι είναι υπέρ ποιοι είναι κατά απορρίπτεται Περνάμε τώρα στην ενοποιημένη 10 του 22. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, Ποχές δεκτή. Ψηφίζουμε τώρα την 381. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ενοποιημένοι 11 στο 23. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ψηφίζουμε τώρα την 400 υπέρ κατά δεκτή. 407 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 149 περιβάλλον υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 408 υπέρ. 408 κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε λοιπόν ηλεκτρονικά την 408 Σμιθ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας δεκτή. 409 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 410 γκέρλινγκ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 411 γκέρλινγκ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Περνάμε τώρα στην 412 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 413 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 414 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ψηφίζουμε τώρα την 415 υπέρ. Κατά. Ε, εντάξει, πρέπει να δώσω Είσαι σίγουρη. Απορρίπτεται. 416 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 416. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 417 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Περνάμε στην 44 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 156. Ποιοι είναι υπέρ. 156 περιβάλλον. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ε, δύο κατά αποχές απορρίπτεται 428 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Περνάμε στην 431 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 158. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 432 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ή μάλλον όχι. Δεκτή διορθώνει ο πρόεδρος. 159 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 160 περιβάλλον συγγνώμη, διορθώνει ο πρόεδρος, 162 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 164 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 165 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 436 υπέρ, Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 436 ψηφίζεται. Πέρασε η ψηφοφορία. Περνάμε στην 4.45. 4.45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 4.45. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζεται. Απερίφθη. Εκατόν εβδομήντα περιβάλλον. Ποιοι είναι υπέρ. Εκατόν Κατά. Δεκτή. 448. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. 171 έμβη υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 450 γέγγελ υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 172 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 451 υπέρ, κατά, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 451. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορίας. Δεκτή. 452 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 453 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 174 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 455 υπέρ κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 455. Ψηφίζουμε. Πέρα της ψηφοφορίας γίνεται δεκτή. 175 περιβάλλον υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος στην 175 ψηφίζουμε. Δεκτή λοιπόν. 4.56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στην 4.58 Λιούπτσεβα. Είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 462 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 463 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 464 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 465 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 466 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 467 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 179 περιβάλλον υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 180 περιβάλλον υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 468 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 469 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα 470 γέγγελ υπέρ κατά αποχές δεκτή και αυτή και οι υπόλοιπε μέσα σε αυτή. 473 Αγιούζο ποιοι είναι υπέρ κατά δεκτή 185 ένβη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 'Πηγαίνουμε λοιπόν στην 480. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 481 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 187 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 483 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 487 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 50 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 490 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την 490 ψηφίζεται Ok, approvato. Adesso andiamo al 492. Andiamo Περνάμε στην 492. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 494 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 498 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 500 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. 501 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 192 ένβη ποιοι είναι υπέρ κατά απορρίπτεται ηλεκτρονικός έλεγχος 192 ψηφίζεται τέλος δεκτή Περνάμε τώρα στη 505 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 506 υπέρ, κατά, δεκτή. 507 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 508 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 509 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 193 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Πηγαίνουμε τώρα στην ομαδική τροπολογία ε ή αγγλικό. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. 194 περιβάλλον. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 195 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Πέντε δεκαεπτά υπέρ κατά αποχές δεκτή. 5.18 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Απορρίπτεται η 5.18. 5.21 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 522 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 524 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 523 υπέρ κατά αποχές. Ο Ζωζέ λέει όχι. Έλεγχος ηλεκτρονικός λοιπόν για την 523. Δεκτή. 5.25 και είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5.28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στην 5.39 του 78. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έλεγχος λοιπόν για την 539, ηλεκτρονικός έλεγχος ψηφίζεται. Γίνεται δεκτή λοιπόν η 539 Κόστιγκερ. 5.40 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 5.42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στην 5.56 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 5.57 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 198 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 199 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 200 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τώρα πηγαίνουμε στην 202 περιβάλλον υπέρ. Υπέρ. Κατά. Απερίφθη. Μετά 566 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 568 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 570 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 205 υπέρ κατά απορρίπτεται. 206 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την 52 ψηφίζεται πέρα στις ψηφοφορίες. γίνεται δεκτή. 53. Τι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 573. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 574 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 576 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 576 παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας γίνεται δεκτή. Ψηφίζουμε τώρα την 577 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 578 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 579 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 211 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 580 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 581 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 582 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 583 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 213 υπέρ κατά απορρίπτεται. 586 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 587 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 215 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 589 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 216 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 217 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 591 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 593 υπέρ. Κάποιος ζητά ηλεκτρονικός έλεγχος για την 591 ψηφίζεται. Πέρα της ψηφοφορίας. «22 υπέρ 20 κατά δεκτή». 594 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 595 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 219 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 596 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 598 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Φτάνουμε μετά τώρα στο κάπα, στην ομαδική κάπα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έξι μηδέν επτά. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εξακόσα οκτώ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 609 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 610 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 611 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ψηφίζουμε τώρα την 224 ένβη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 615 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Α. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 615. Πέρα της ψηφοφορίας. 28 υπέρ, 12 κατά. 628. Αγιούζο υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 225 NV υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. ομαδική F αγγλικό υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ψηφίζουμε λοιπόν την 636 υπέρ κατά δεκτή. Έξι τριάντα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 6.37. Α, όχι. 6.38. Σμιτ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έξι υπέρ κατά αποχές Δεκτή. 234 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 234 ψηφίζεται. Δεκτή. 6.44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6.47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 236 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 648 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες. Η 648 γίνεται δεκτή. 649 υπέρ. Κατά. Απερίφθη. 650. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απερίφθη. 651 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 652 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Περνάμε τώρα στο G αγγλικό υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές. 654 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 6.55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6.57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Α, έχω κάνει κάποιο λάθος λέει ο πρόεδρος. Γίνεται δεκτή η 657. 54 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 659 μπαράτσου υπέρ κατά αποχές δεκτή. 660 υπέρ κατά. Ε, πρέπει να υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος για την 660. δεκτή. Ψηφίζουμε τώρα την 662. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 664 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 243 περιβάλλον. υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 243 παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Δεκτή τελικά. 55 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 665 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 244 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 245 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 671 υπέρ κατά Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο για την 671. Ψηφίζετε. Πράγματι 23 υπέρ 17 κατά. Ψηφίζουμε τώρα την 674 υπέρ. Κατά. 246 περιβάλλον υπέρ κατά αποχές και εδώ είναι δύσκολο να κρίνεις ψηφίζουμε ηλεκτρονικά λοιπόν για την 246 απερίφθη με μία ψήφο διαφορά. 6.75 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 6.76 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 6.77 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 6.78 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 6.79 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 680 ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Κάνουμε ένα μικρό άλμα, πηγαίνουμε στην 253 περιβάλλον, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη, 254 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 688 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 690 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 692 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 696 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Συμβιβαστική υπαριθμών 3. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τώρα ψηφίζουμε την 706 Γκέρλινγκ υπέρ κατά αποχές απερίφθη 707 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 708 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 710 υπέρ κατά αποχές δεκτή ομαδική ήτα H αγγλικό 1 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή 714 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται θα γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος για την 714 άρχεται η ψηφοφορία Πέρα τη ψηφοφορίας. Δεκτή. Δεκτή. Εφτά δεκαπέντε. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 716 υπέρ κατά αποχές υπέρ. 259 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 717 μπαράτσου υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 718 υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. 719 υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. 29 αλία υπέρ κατά αποχές δεκτή. 30 αλία υπέρ κατά αποχές δεκτή. 720 υπέρ κατά απερίφθη νομίζω 721 υπέρ κατά απερίφθη 722 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Στο H2 λοιπόν ή τα δύο ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. 723 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 724 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 725 υπέρ κατά αποχές δεκτή 726 υπέρ κατά αποχές απερίφθεια 727 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 728 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 729 υπέρ κατά αποχές απερίφη. Ηλεκτρονική ψήφος για την 729. Ελέγχουμε. 729. Γίνεται δεκτή. Μεγάλη πλειοψηφία. Ψηφίζουμε τώρα την 730 Γκέρλινγκ Νίκολσον υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τώρα 731 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 732 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2.63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την 733 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα την 735 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 737 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 267 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 268 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 739 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 742 υπέρ κατά αποχές δεκτή 270 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 60 εισηγητής υπέρ κατά αποχές δεκτή Ψηφίζουμε τώρα την 745 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Την 61 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Την 273 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Την 749 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Την 750 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Την 62 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 751 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 752 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 753 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 760 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 275 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Περνάμε τώρα ε, στο I, στο Ι, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτό. 281 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 64 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 779 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Πηγαίνουμε λοιπόν σε αιτιολογικές σκέψεις. 2. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 70. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 71. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 73. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρι... δεκτή. 3. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τέσσερα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τρία υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ένα αλία υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την ένα αλίας. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Εβδομήντα πέντε υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εβδομήντα έξι υπέρ κατά αποχές δεκτή 77 υπέρ κατά αποχές δεκτή θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο για την 77 άρχεται η ψηφοφορία 77 Westlund ed approvato. Δεκτή. Επτά υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Οκτώ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Εβδομήντα οκτώ υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. εννέα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 81 υπέρ κατά δεκτή. 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 12 περιβάλλον υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 13 περιβάλλον υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 84 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. 15 περιβάλλον υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 17 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 86 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή.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 Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 92 ψηφίζεται. Πέραστη ψηφοφορία απερίφθη. Ψηφίζουμε τώρα την 94 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 25 περιβάλλον υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 101 λιούψεβα. υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 102 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 103 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 30 περιβάλλον υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 105 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 106 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 107 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 112 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 113 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 114 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 115 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Απερίφθη, απερίφθη 116 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 117 λιούψεβα υπέρ, Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 38 περιβάλλον. Υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 121. Υπέρ. Κατά. Αποχές. φορά. 122. Απορρίπτεται. 124 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 126 γκέβλεν υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Περιβάλλον 42 υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 42. Ψηφίζεται. Δεκτή. Η 42. 128 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 129 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 130 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 44 περιβάλλον υπέρ κατά αποχές περιβα... Ε, απορρίπτεται. 131 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 6 όχι. 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 133 υπέρ κατά αποχές δεκτή η 133. 46 περιβάλλον, ή όχι, 47 μάλλον περιβάλλον, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 134 υπέρ, κατά. 135 ματιό υπέρ, κατά. Αποχές, απερίφθη θα έλεγα. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Για την 135 ελέγχουμε, ψηφίζεται. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί λέει ο πρόεδρος. Όχι, έγινε δεκτή τελικά. Ο Ντέις έχει δίκιο. 7 του εισηγητή. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 136 Βέσλοντ, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 48 περιβάλλον, υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 49 περιβάλλον, υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 50 περιβάλλον, υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Ψηφίζουμε τώρα με την 138 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 52 ε, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 53 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 54 περιβάλλον υπέρ, κατά, Δεκτή. 55 περιβάλλον υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 139 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 58 περιβάλλον υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 59 περιβάλλον υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. 60 περιβάλλον υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 142 ή μάλλον 100 α, 62 υπέρ κατά απερίφθη. 64 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 147 Στάντλερ υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 148 Στάντλερ υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Τώρα λοιπόν ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για το σύνολο της νομοθετικής προτάσεως όπως τροπολογήθηκε. Ξεκινάτε την ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. δεκτή και τελευταία ψηφοφορία για σήμερα πρόταση νομοθετικού ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. Καλώς. Συγχαρητήρια λοιπόν. Κάναμε πραγματικά μια κουραστική ψηφοφορία. Θα διακόψουμε για λίγα λεπτά και θα ξεκινήσουμε μετά με το σημείο 8. Έχουμε ξανά ψηφοφορίες για τα προληπτικά μέτρα για τα ζυζάνια. Un Presidente, votiamo. Pronti. Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι. Iniziamo. ξεκινάμε. Συνάδελφοι, ξεκινάμε με τη δεύτερη περίοδο ψηφοφοριών, το 8. Σημείο 8 στην ημερήσια διάταξη. Σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης λοιπόν. Πρόταση για τους επιβλαβείς οργανισμούς των φυτών. Έχουμε τον εισηγητή μας ε, και Φαϊμόνα που έχει καθίσει. Έχουμε πολλές τροπολογίες. <clears throat> Δεν θα είναι τόσο μακρόχρονη ψηφοφορία όπως η προηγούμενη, αλλά χρειάζεται λίγη υπομονή, χρειάζεται κάποιος χρόνος. Και ο εισηγητής ε, θέλει ίσως να λάβει τον λόγο. Παρακαλώ, Ινέκ. Θέλεις να παρέμβεις. Ευχαριστώ πολύ σύντομα πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το λόγο να παρέμβω. Έχουμε σχεδόν 500 τροπολογίες που κατατέθηκαν και πιστεύω ότι όλοι γνωρίζουμε <clears throat> ποια είναι τα ουσιοδέστερα σημεία σε αυτό το θέμα και περί τίνος πρόκειται ουσιαστικά. Αυτό που πρέπει να κάνουμε λοιπόν είναι να ψηφίσουμε την πρόταση. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε διανατάσεω των, σειρών, ε, των χειρών, εκτός αν υπάρχουν αμφιβολίες, οπότε θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Είμαστε έτοιμοι. Ξεκινάμε λοιπόν. Ξεκινάμε. Λοιπόν, Φύγαμε. Άρθρο 1. Τροπολογία 66. Ντάνσιλα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 67. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 68. Άγκο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 70. Σαντεμόζε υπέρ. Κατά Αποχές απορρίφθηκε. Εντάξει, απορρίφθηκε. Τροπολογία 10, εισηγή του υπέρ. Κατά, αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 69, Ανδρίο υπέρ. Κατά, αποχές απορρίφθηκε. 71, Ανδρίο υπέρ. Κατά, αποχές απορρίφθηκε. 72, Γέγκλε υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 73 γέγλε υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 75 γέγλε υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 77 γέγλε υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε. 78 Χόισλινγκ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 79 Χόισλινγκ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 80 Νίκολσον υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε το, την τροπολογία 80. Άρχεται, ψηφίζουμε την 80 Νίκολσον. Ψηφίσατε όλοι. Απορρίφθηκε. Συνεχίζουμε. Ψηφίζουμε διανατάσεως των χειρών. 81. Χόισλινγκ υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 82 Χόισλιν υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 83 83 Ντελάνγκε υπέρ κατά αποχές αεγκρίθηκε 84 Ντελάνγκ υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 85 Ντελάνγκ υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. NV27 υπέρ κατά Θα λέγα απορρίφθηκε. Εντάξει, απορρίφθηκε. 88 ένβη υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 89 Χόισλινγκ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 90 Ντάνσιλα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 91 ένβη υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 92 Ντάνσιλα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 93 Χόισλινγκ υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε NV30 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε πάμε τώρα στην 95 Ντάνσιλα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 96 Χόισλινγκ υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Από κοινού NV31 και 32 υπέρ αυτών. Κατά αποχές απορρίφθηκαν. Τώρα θα πάμε στην 99 Γκαρσία Πέρες και άλλων. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Ένβη 33. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Ένβη 34. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 103 Γκαρσία Πέρες υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 105 Αγιούσο υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Ένβη 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Ένβη 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 111 Μακίνταρ υπέρ κατά απόχες απορρίφθηκε 112 γιούσο υπέρ κατά απόχες εγκρίθηκε μου είπαν ότι περάσαμε ένα άρθρο και πρέπει να το ψηφίσουμε είναι το 94 αντάνσιλα 94 λοιπόν 94 υπέρ κατά απόχες απορρίφθηκε Το 94 εγκρίθηκε, λέτε. Ε, συγγνώμη, ωραία. Να σηκώνετε τα χέρια. Ψηφίζουμε την τροπολογία 94 Ντάντσιλα, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε λοιπόν. Ε, όταν λέμε εγκρίθηκε, εγκρίθηκε. Τώρα συνεχίζουμε με τον κατάλογο ψηφοφορίας. Εντάξει, πάμε στην 114. Αγιούσο, υπέρ. Κατά αποχές, εγκρίθηκε. NV39. Όχι, εντάξει, έχουμε πιο πριν την 11 του εισηγητή. Μετά από αυτήν, υπέρ. Κατά αποχές, εγκρίθηκε. 116 γκίρλινγκ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. NV41 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. NV42 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Εκατόν Μακριντάρ υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 12 εισηγητού υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. NV43 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Εντάξει, να ελέγξουμε. Ελέγχουμε. Ψηφίζουμε τη 43 NV ηλεκτρονικά. Άρχεται. Απορρίφθηκε με μία ψηφοδιαφορά. Απορρίφθηκε. Πάμε τώρα στην 126 Νίκολσον υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 127 Χόισλινγκ υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Ένβη 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 128 Νίκολσον όχι 129 129 συγγνώμη Νίκολσον υπέρ όχι, δεν θα ψηφιστεί. Ωραία, πολύ καλά. Πάμε στην 45, ένβη, εντάξει. Α, πρέπει να τις ψηφίσουμε αυτές. Ωραία, ψηφίζουμε ομού 129, 130, 131, υπέρ αυτών. Κατά. Είναι ομαδική ψηφοφορία ομού 129, 130, 131 από κοινού. Με μία ψηφοφορία. Εντάξει, 129, 130, 131. Υπέρ αυτών. Κατά. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 129, 130, 131. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. <clears throat> Απορρίφθηκαν. Ωραία. Λοιπόν, Πάμε τώρα στην NV45 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 132 Χόισλινγκ υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. NV46 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. NV47 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. 133 Αντρίο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 134 Χόισλινγκ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. NV48 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. NV49 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 135 Χόισλινγκ υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. 136 Νίκολσον υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 137 Νίκολσον υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 138 Ράιμερς υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 139 Ράιμερση και άλλων υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 142 Μπρίτα Ρέιμερς υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 143 Χόισλινγκ υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε NV 53 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε NV54 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 14 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 144 ντελάνχ υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε NV56 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 145 χόσλινγκ υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 146 χόσλινγκ υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 147 Ρέιμερς υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε NV57 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Εγκρίθηκε λέτε. Ωραία. Ζητώ συγγνώμη. NV57 υπέρ. Μάλιστα. Ωραία. Κατά αποχές εγκρίθηκε η 57. Εγκρίθηκε. Πάμε στην 148 Ντελάγκα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. NV58 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. NV150 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Ένβη 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 153 ντάνσιλα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Ένβη 61 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 154 Χόισλινγκ υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 155 Ντελάνκ υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 156 Γκαρσία Πέρες υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 158 Γκαρσία Πέρες υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 160 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 162 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 164 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 166 Χόισλινγκ υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 64 υπέρ κατά απόχες εγκρίθηκε 169 σαρντεμόζε υπέρ κατά απόχες απορρίφθηκε 170 χόισλινγκ υπέρ κατά απόχες απορρίφθηκε 165 υπέρ κατά Αποχέ, απορρίφθηκε 171 χόισλινγκ υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 16 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 17 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 172 Φράνκο Ανδριό υπέρ 172. Α, εγκρίθηκε. Ωραία. 174 Αγιούσο λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. Και τώρα θα πάμε στην ένβη 67 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. Ένβη 68 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 169. 69 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε έτσι, ωραία. 18 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 176 Ανδρέα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 177 Χόισλινγκ υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 178 Αγιούσο υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Ένβη 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 182 Αγιούσο υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 184 γκαρσια Πέρε Πέρες υπέρ Αποχέ. αποχές Ένβι NV74 υπέρ κατά Αποχέ. εγκρίθηκε η 187 Ρέιμε. υπέρ κατά Αποχέ. εγκρίθηκε η 19 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 188 Αγιούσο υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 20 του υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η α υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Θα ελέγξουμε λοιπόν. Ψηφίζουμε την παγιωμένη τροπολογία Α. Α. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Και απορρίφθηκε. Λοιπόν, πράγματι απορρίφθηκε. 19 <clears throat> υπέρ 22 εναντίον. Η α, απο, η α λοιπόν απορρίφθηκε. Και τώρα περνάμε στην 189 Ανδρέα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Και περνάμε στον μπλόκο ομάδα τροπολογιών Ανδρέα υπέρ αυτών. Κατά αποχές εγκρίθηκαν οι τροπολογίες του μπλοκ αυτού. Αντριέ. Περνάμε στην 197 γουτιέρες υπέρ, κατά, αποχές. Λοιπόν, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά, ασαφές το αποτέλεσμα. Άρχεται η ψηφοφορία, 197 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας για την 197 που απορρίφθηκε. Πάμε στην 199. Γκαρσία Πέρες. Υπέρ. Όχι, έτσι, όχι. Ωραία. Η 200 τώρα. 200. Αγιούσο. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά θέλετε. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την τροπολογία 200 Αγιούσο. Πέρας ψηφοφορίας και απορρίφθηκε με μία ψήφο διαφορά, 21 εναντίον 20 υπέρ, απορρίφθηκε. 201, Γκασία Πέρες, διανατάσεως του, διακόπτει ο πρόεδρος. Συγγνώμη ζητώ. Λοιπόν, είχαμε μια ψηφο διαφορα 21 εναντιον 20 υπερ απορριφθηκε 201 αγκασια περες διανατασεως το διακοπτει ο προεδρος συγγνωμη ζητω λοιπον ειχαμε μια δυσκολια 212, Αγιούσο, υπέρ, διανατάσεως, 212 λοιπόν, υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. 214 Χόισλινγκ υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 215 Γασία Πέρες υπέρ κατά απορρίφθηκε. 217 Αγιούσο υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 219 Γασία Πέρες υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 221 Χόισλινγκ υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 21 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 222 Γασία Πέρες υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 22 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 225. για Πέρεση. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Να ελέγξουμε λέτε. 225 λοιπόν ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. «225 λοιπόν, έτσι, 225 ηλεκτρονικά, άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας ε, για την 225 εγκρίθηκε λοιπόν με μεγάλη πλειοψηφία. 227 διανατάσεως Γκαρσία Πέρες 227 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 231 Αγιούσο υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Περνάμε στην τροπολογία, παγιωμένη τροπολογία B, Β, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Περνάμε στην ενσωματωμένη τροπολογία C, Γ, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 241, Αγιούσο, υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 242 Σαλτεμόζε υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 243 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 23 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 244 Ανδρέο υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 245 δελάνκ υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 24 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 248 Νίκολσον υπέρ. Όχι, όχι. Εντάξει αποσύρθηκε αυτή. Μάλιστα. 25 του εισηγητή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 249 Νίκολσον υπέρ κατά εγκρίθηκε 251 Χόισλινγκ υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 252 Χόισλινγκ υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 253 Χόισλινγκ υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 254 Χόισλινγκ υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. 255 Χόισλινγκ υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. 258 Αντριο υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Να ελέγξουμε λέτε. Ωραία. Ελέγχουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 258 Ανδριού Άρχεται η ψηφοφορία. Μάλιστα. Πέρας ψηφοφορίας. Και απορρίφθηκε. Μάλιστα. 256 Χόισλινγκ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 257 Σάλτεμοζε υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. 259 Ανδριέ υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 26 εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 261 Χώστιν υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 27 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 200 πως είπατε εσείς για το 27 θέλετε να ελέγξουμε. 262 λοιπόν, Χόισλινγκ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 28 του συγητή υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 263 Χόισλινγκ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 264 υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. 265 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 266 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 267 Ανδρείο υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. NV79 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 268 Σιλβέστρης υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Ένβι 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 270 Ιούσο υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 271 Γασία Πέρες υπέρ κατά απορρίφθηκε. 273 Μακιντάρι υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 274 Χόισλινγκ υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 275 Χόισλινγκ υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε Ένβι 81 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 29 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 276 Χόισλινγκ υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 277 Χόισλινγκ υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 278 Ντελάγκε υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 279 Νίκολσον υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 280 Γκίρλινγκ υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 30 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. NV82 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. NV83 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Του εισηγητή 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 84 NV υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Η 32 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Ένβιο 85 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 33 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Η 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε θα λέγα έτσι ωραία 282 Νίκολσον υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 283 Νίκολσον υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 285 τελάνε υπερ υπέρ κατά αποχές 187 NV87 υπέρ όχι συγγνώμη εντάξει 286 286 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 280 288, 288 Ιούσο υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 289 Αγιούσο υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Περιβάλλουν 90, απορρίπτεται. 290 Αγιούσο υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. 291 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. 292 υπέρ, κατά, αποχές δεκτό. 293 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 92 περιβάλλον υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Περιβάλλον 93 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Περιβάλλον 94 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Περιβάλλον 95 υπέρ, κατά, αποχές δεκ, απορρίπτεται. 96 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 97 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 98 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 34 εισηγητή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.94 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.96 υπέρ κατά αποχές δεκτή 299 υπέρ κατά αποχές δεκτή Χάουσλινγκ 301 υπέρ κατά αποχές δεκτή απορρίπτεται μάλλον 302 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 303 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 304 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 305 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 306 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 307 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 308 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 309 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Περιβάλλον 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 310 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 313 τώρα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Δεν έχει πολύ τύχη ο Χόλσλινγκ σήμερα, λέει ο Πρόεδρος. 3.14 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 3.15 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Περιβάλλον 104 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 316 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 317 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 318 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 319 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 320 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 321 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 322 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 323 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 324 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 325 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 326 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 327 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 328 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 329 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 330 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 331 υπέρ κατά αποχές δεκτό. δεκτό 108 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στις αιτιολογικές σκέψεις. Περιβάλλον 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 36 Χάουσλινγκ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. NV2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 37 η MV3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο για την τροπολογία 37. Πέρα τη ψηφοφορίας. Απερίφθη. Φτάσαμε τώρα στην 38. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 39. Υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 40. Υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Περιβάλλον 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 1 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και εγώ αναρωτιόμουν αν υπάρχουν συμβιβαστικές αλλά δεν υπάρχουν λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν 7 απορρίπτεται. 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ένβι, 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 45 Χόισλινγκ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2 εισηγητή, υπέρ, κατά, αποχές, ΕΝΒΙ NV10, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 47 Χόισλινγκ, υπέρ, κατά, υπέρ, απορρίπτεται. 11 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 48 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 50 Κοιτάξτε, θα γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 3 του εισηγητή. Εντυρέει direi che Νομίζω ότι έχει γίνει δεκτή, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Ομόφωνα έχει <laughs> γίνει δεκτή. Ποιος το ζήτησε να το ψηφίσουμε. Νομίζω ότι το πετύχαμε. 50. Ο Άγνιου έχει ζητήσει το λόγο. Μετά από την ψηφοφορία αυτή επιμένω για αυτόν ο οποίος ζήτησε τον έλεγχο να σηκώσει το χέρι του να τον δούμε. <laughs> Καλώς, έχετε δίκιο κύριε Αγνιού. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία της 50 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 51 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 52 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Περιβάλλον 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Εισηγητής 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 54 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ένβη 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 58 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Πηγαίνουμε τώρα στο περιβάλλον 17 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 6 εισηγητής υπέρ κατά αποχέ δεκτή. 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 18 περιβάλλον υπέρ κατά αποχές δεκτή. 19 περιβάλλον υπέρ κατά αποχές δεκτή. 20 περιβάλλον υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 21 περιβάλλον υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές δεκτή. 9 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές δεκτή. Περιβάλλον 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 60 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Λοιπόν τώρα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την νομοθετική πρόταση όπως έχει τροπολογηθεί. Ψηφίζεται ηλεκτρονικά. E Δεκτή και στο τέλος ψηφίζουμε το νομοθετικό ψήφισμα, την πρόταση νομοθετικού ψηφίσματος. Ψηφίζουμε. Λοιπόν τελειώσαμε. Ευχαριστούμε τον εισηγητή και συγχαίρουμε τον εισηγητή. Αυτό είναι το αποτέλεσμα.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 παραγωγή και διάθεση στην αγορά αναπαραγωγικού φυτικής προέλευσης υλικού. Η είναι ο Σερτζο Πάολο Φραντσέσκο Σιλβέστρης. Περνάμε λοιπόν στην ψηφοφορία στην πρόταση της Επιτροπής. Όπως όλοι οι ενθυμίστε, συνάδελφοι, είχαμε συζητήσει το θέμα αυτό επανειλημμένα είχαν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα από αυτή την ομοθετική πρόταση και στην τελευταία συνάντηση των συντονιστών είχαμε πει ότι θα απορρίψουμε. Ε, πρώτα θα ψηφίσουμε λοιπόν την τροπολογία απόρριψης της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά στην ομοθετική πρόταση. Και μετά πάλι τίποτα. Λοιπόν όπως είπα προτείνω να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά ψηφίζουμε λοιπόν συνάδελφοι την ε, τροπολογία 91 με 98 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. 91 e 98 che sono identici, vero? Sì, sì, sì. Ok. chiusa la... 91-98 είναι ταυτόσιμες. Τέλος της ψηφοφορίας. Έχουμε μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία, 37 υπέρ, 2 κατά. Καμία αποχή. adesso, adesso votiamo. Τώρα πλέον θα ψηφίσουμε την πρόταση νομοθετικού ψηφίσματος για την απόρριψη. Άρχεται η ψηφοφορία. Votazione chiusa. Τέλος της ψηφοφορίας. Το ίδιο αποτέλεσμα, 37 υπέρ, 0 ε, ε, αποχές μάλλον και 2 κατά. Καλώς συνάδελφοι, σε αυτή τη φάση πλέον Sì. Adesso dobbiamo votare invece. Θα πρέπει να ψηφίσουμε το κείμενο για την προφορική ερώτηση, πάντα ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για την προφορική ερώτηση. Chiusa la votazione. Πέραση ψηφοφορίας. Έχουμε λοιπόν το αποτέλεσμα 34 υπέρ, 3 κατά, 1 αποχή. Μεγάλη πλειοψηφία λοιπόν και για την προφορική ερώτηση. Ο Ζωζέ Μποβέ έχει ζητήσει το λόγο. Θεωρώ ότι στο κείμενο βλέπω ότι υπάρχουν δύο σημεία που λείπουν και θα έπρεπε, κατά σημαντικά και θα πρέπει να αναφέρονται. Πρώτον, η αναφορά παραπομπή στην σύμβαση για την ε, βιολογική βιοπικιλότητα που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει οπωσδήποτε αυτό το κείμενο να αναφέρεται. Και δεύτερον, να πρέπει και πάλι να ξεκαθαρίσουμε ρητός ε, την ανταπόκρισή μας ε, στην βιοποικιλότητα για ε, τα δικαιώματα των καλλιεργητών. Εάν δεν έχουμε αυτά τα στοιχεία, νομίζω ότι το ζήτημα που θέτουμε προς την Επιτροπή δεν θα είναι ορθό. Και αν δεν κάνουμε αυτό, πρέπει να κινηθούμε προς άλλα κείμενα που προτείνουν οι πολιτικές ομάδες. Κατά τη γνώμη αυτό θα ήταν λάθος, Μένω λοιπόν εδώ είναι πολύ πιο σωστό και θα είναι πολύ καλύτερο μήνυμα προς ε, την Επιτροπή. Okay. Ευχαριστώ Ζωζέ. Θα ήθελα να να διευκρινίσω ότι μιλάμε για την προφορική ερώτηση. Ψηφίσαμε την προφορική ερώτηση, την αρχική δεν υπήρχε αμφιβολία, αλλά θα πρέπει, έχουμε αμφιβολίες για το συγκεκριμένο ψήφισμα και τα σημεία αυτά θα τα επεξεργαστούν οι πολιτικές ομάδες όπως το έθεσαν και οι πράσινοι και θα περάσουν μετά στην ψηφοφορία, στην Ολομέλεια πια. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο. Δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλος το λόγο. Θα συνεχίσουμε λοιπόν όπως είχαμε αποφασίσει. Περνάμε τώρα στο σημείο 10 της ημερησίας διάταξης διαχείριση των δαπανών των σχετικών με την τροφιμική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των διαλόγων και έγκριση του ενοποιημένου κειμένου. Θα δώσω το λόγο στην συνάδελφο Ανιές Λεμπρά για να μας παρουσιάσει τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων. Έχετε το λόγο κυρία Λεμπρά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το κείμενο που υποβάλλουμε σήμερα συμπεριλαμβάνει τα βασικά αιτήματα του Κοινοβουλίου σε τέσσερα σημεία. Αφενός έχουμε την προσφυγή μας στα ε, αντίστοιχα κονδύλια. Δεν υπάρχουν πλέον κίνδυνοι για τις πληρωμές του γεωργούς και σε περίπτωση έλλειψης ε, κονδυλίων ε, στη γραμμή του προπολογισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ε, προσφύγει σε μέσα ευελιξίας για να καλύψει τον προπολογισμό. Δεύτερον, ε, δεύτερο σημείο διαπραγματεύση είναι ο κατάλογος των επιζώτιων που έχουν ενσωματωθεί στην ε, βασική πράξη μέσω παραρτήματος για να γίνει πιο ευανάγνωστο το κείμενο αλλά και για να υπάρχει μεγαλύτερο έλεγχο από το Κοινοβούλιο. Το τρίτο σημείο είναι ο κατάλογο ε, των επιλέξιμων δαπανών. Δεν θεωρούμε ότι έχει εμπλουτιστεί επαρκώ. Και τέλος ε, προσθέθηκαν ε, σημεία τα οποία είχαν παραλυφθεί ας πούμε από την Επιτροπή. Και τέταρτο σημείο, ζητήσαμε το Κοινοβούλιο να συμπεριληφθεί μέσω κάτεξοδότησης πράξεων στο στην ε, διαμόρφωση του προγράμματος εργασίας. Είναι δύσκολο αυτό να εφαρμοστεί στην πράξη, γι' αυτό ενισχύσαμε τελικά ε, την βασική πράξη, τον ίδιο τον κανονισμό. Με αυτόν τον τρόπο το Κοινοβούλιο συμμετέχει στον ορισμό ε, των πολιτικών προτεραιοτήτων και η Επιτροπή διατηρεί την ευελιξία που χρειάζεται για να εκπαιδεύσει μια κατάλληλη πολιτική. Σε αυτά τα τέσσερα σημεία λοιπόν ε, έγιναν σεβαστές οι απόψεις μας και αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εκπροσώπους και του Συμβουλίου και της Επιτροπής με τους οποίους ε, ε, εργαστήκαμε από κοινού και με πολύ καλό τρόπο κατά τη γνώμη μου και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερως τη Γραμματεία Άγκρη και τους σκιώδεις συζητητές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Λεμπρά. Τώρα θα πρέπει να ψηφίσουμε για ανατάσσεως χειρών. Α, όχι, ηλεκτρονικά. Θα πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, λέει ο Πρόεδρος, για τις ενοποιημένες τροπολογίες που μας παρουσίασε η κυρία Λεμπρά. Ψηφίζουμε. Πέρα της Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Θα συνεχίσουμε λοιπόν. Δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλος το λόγο και περνάμε στο σημείο 11, τροποποίηση του κανονισμού 1166 σχετικά με τις έρευνες για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όσον αφορά το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2018. Εγώ είμαι ουσιαστικά ο εισηγητής. Θα πρέπει και εδώ να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία. Ο κανονισμός μας δίνει τη νομική βάση. Αυτή τη στιγμή οι έρευνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό εντάσσονται σε δύο περιόδους του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και δεν μπορέσαμε έτσι ταυτόχρονα να καθορίσουμε το ύψος χρηματοδότησής τους. Πρέπει λοιπόν να ψηφίσουμε την πρόταση για να διασφαλίσουμε την λειτουργία των ερευνών αυτών, έτσι ώστε να συνεχιστούν κατά τη διάρκεια και του νέου πολιετούς δημοσιονομικού απαιτείται με ταχύτητα η υιοθέτηση της πρότασης αυτής για να μην υπάρξει καθυστέρηση στην ανάπτυξη της βάσης δεδομένων και στην προπαρασκευή των μέτρων συγχρηματοδότησης και να μην καθυστερήσουν και οι επόμενες μελέτες, έρευνες που θα πρέπει να ξεκινήσουν το 2016. Το Συμβούλιο είπε ότι θα εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής χωρίς τροποποίηση Απαιτείται λοιπόν και από πλευράς μας και από το Συμβούλιο να προχωρήσουμε με ταχύτητα. Λοιπόν δεν ξέρω αν υπάρχουν παρατηρήσεις, νομίζω ότι μπορούμε να ψηφίσουμε απευθείας ηλεκτρονικά και σε αυτή την περίπτωση. Είστε όλοι υπέρ. Πέραση ψηφοφορίας. πολύ μεγάλη πλειοψηφία, ένας μόνο ψήφισε κατά και έχουμε μία ψήφο αποχής. Και πηγαίνουμε στο σημείο 12 τώρα, όπως γνωρίζετε συνάδελφοι, υπάρχει μία προφορική ερώτηση επί τη βάση του άρθρου 115 που αφορά την Διεθνή Έκθεση του Μιλάνου το 2015. Πρόκειται για μια σημαντική ευκαιρία για όλη την Ευρώπη και όχι μόνο για την συγκεκριμένη χώρα είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο μας αφορά και σαν Επιτροπή Γεωργίας αναμένονται 20 εκατομμύρια επισκεπτών σημαντική ευκαιρία για την ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών σε τομείς όπως η τροφιμική ασφάλεια, η αηφορία. Τα θέματα λοιπόν της εκθέσεως αυτής εντάσσονται και στον αγροτικό και τροφιμικό τομέα και θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λίγο εμείς σε τι επίπεδο θα βρίσκονται τα μηνύματα που θα μεταφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και γι' αυτό καταθέσαμε μια προφορική ερώτηση για να ακολουθήσει συζήτηση στην Ολομέλεια. Λοιπόν, ελπίζω να το πετύχουμε στις επόμενες ε, ολομέλειες του Στρασβούργου πριν το τέλος της κοινοβουλευτικής περίοδου. Συμφωνούμε όλοι λοιπόν, θεωρείτε δεκτή η πρόταση αυτή. Δεν χρειάζεται ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία, σας ευχαριστώ. Δεν έχουμε κάτι άλλο για σήμερα. Η επόμενη συνεδρίαση είναι σήμερα το απόγευμα ε, και οι ακροάσεις τις οποίες έχουμε. Ήμασταν λίγο κουραστικοί αλλά σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας. Θα τα πούμε το απόγευμα στις 3 το μεσημέρι.